seats. We're about to begin the votes. Δείτε συνάδελφοι, γιατί αρχίζουν οι ψηφοφορίε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συνοπτικά πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Αν όχι, τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και όποιος δεν κάθεται δεν θα ψηφίζει. παρακαλώ. The Kaiser. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επανέλθω σε ένα θλιβερό γεγονός που εξελίχθηκε χθε εδώ μέσα στην Ολομέλεια που είναι ε, ανάξιο του Κοινοβουλίου. Προσβλήθηκε ο κύριος Ερμάν Βονροπέ, πρόεδρος του Συμβουλίου. Βέβαια μπορεί να αμυνθεί μόνος του. Μπορεί. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου είναι σε θέση να αμυνθεί. Αλλά δεν δέχομαι εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο οποιοδήποτε να πει για τη χώρα μου ότι δεν είναι χώρα. Είναι μια χώρα ιδρυτικό μέλος της Ένωσης που σύντομα θα έχει την Προεδρία και δεν καταλαβαίνω πώς εδώ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους ε, προφορικές μεθόδους και απαιτώ συγγνώμη. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης της κυρίας Βαλεάν σχετικά με την ανακοίνωση στην Επιτροπή των Επενδυτικών Σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπάτεν έχει το λόγο on a point of order. Thank you. Point of order, Mr. President. I'd like... Διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω υπό τον ίδιο κανόνα που όσοι και η κυρία που μίλησε τώρα και αναφέρθηκε στον άδελφο Νάζελ Φένελτζε. Εσείς μας ε, υποχρέωσαν να πάρουμε τι συνθήκε Λισαβόνη και όταν ο συνάδελφο λέει κάτι, όλοι δεν του αρέσει και διαμαρτυρώνουν. Αυτό είναι πολιτική. Πολιτική έχουμε στη χώρα μα Λοιπόν, θα πρέπει να μάθετε να ακούτε και άλλε γνώμε από εκείνου που σα αρέσουν. Η περισμένη δήλωση ήταν δήλωση απάντηση σε κάτι που λέχθη χθε. Αυτό ήταν ο κανόνα με τον οποίο ήταν, δεν ήταν διαδικαστικό. Το δικαιωτικό σα ήταν εκτό το πιο χρόνο. Περνάμε στην ψηφοφορία τώρα. Προβλέπει την ψηφοφορία επί τη έκθεση κυρία Βαλεάν σχετικά με την ανακοίνωση στην Επιτροπή των Επενδυτικών.